Υποθέσεων μας ανακοίνωσε μία διόρθωση, διόρθωση κάποιων σφαλμάτων σε σχέση με το κείμενο το οποίο εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο. Η διόρθωση αυτή, το διορθωτικό, είναι στο